ευχαριστώ τους κύριους και τις κύριες βουλευτές που έφεσαν τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τελείωσε η συζήτηση. Θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας και πάλι αύριο το πρωί στις 8.30. Καλό σας βράδυ.